Έχετε τις κάρτες ψηφοφορίας μαζί σας, έτσι. Για βρείτε τες. Ωραία. Περνάμε στην ψηφοφορία για την έκθεση όσον αφορά την εφαρμογή της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων στις χώρες μέλη. Η συγγήτρια είναι η κυρία Μπλινκεβιτσούτε και αρχίζουμε την ψηφοφορία. Τροπολογία 36. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 37. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 38 υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι εγκρίνεται, αλλά καλύτερα να λέξουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ. Ψηφίστε ηλεκτρονικά. Πέρας της φοφορίας Εγκρίθηκε. Κυρία Μακάβεν, υπερψηφίσατε, έτσι. Ναι, ναι, ναι, εγκρίθηκε. Τροπολογία 39 τώρα. Εδώ πέρα υπάρχει μια τεχνική προφορική τροποποίηση. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 40. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Να ελέγξουμε. Ωραία. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά για την τροπολογία 40. Μπορείτε να ψηφίσετε. Ε, ψηφίστε παρακαλώ. Πέρα στις φοφορίες. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 41 με προφορική τροποποίηση. Υπάρχουν αντιρρήσεις παρακαλώ στην προφορική τροποποίηση. Όχι, υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 42 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 43 με τεχνική προφορική τροποποίηση υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 44 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 45 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 46 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβιβαστική τροπολογία 3 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 51 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 4 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 58 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 56 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 60 υπέρ, κατά, αποχές, θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Μπορείτε να ψηφίσετε για την τροπολογία 60. Ψηφίστε πέρα τη ψηφοφορίες. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 61 τώρα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 62 υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά για την τροπολογία 62. Μπορείτε να ψηφίσετε πέρα τη ψηφοφορία. Απορρίφθηκε. 63 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 64 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 65 υπέρ, κατά, αποχές, να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Εγκρίθηκε. 66 υπέρ. Τροπολογία 66 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφέ το αποτέλεσμα. Πρέπει να ελέγξουμε ηλεκτρονικά για την τροπολογία 66. Ψηφίστε παρακαλώ. Amendment 66. 66 είπαμε. Πέρας της φοφορίας εγκρίθηκε. Τροπολογία 67 υπέρ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 68 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε ηλεκτρονικά για την τροπολογία 68. Μπορείτε να ψηφίσετε. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 69 με τεχνική προφορική τροποποίηση υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 70 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 71 με τεχνική προφορική τροποποίηση υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική αριθμός 1 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 19 υπέρ,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 αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 2 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 30 σε δύο τμήματα. Θα ψηφίσουμε πρώτα το δεύτερο τμήμα. Υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. δεν χρειάζεται να ψηφίσουμε το πρώτο τμήμα, καταπίπτει. Και πάμε στην τροπολογία 31, υπέρ, κατά, αποχές, να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Τροπολογία 31. Ψηφίστε. Πέρα στις φοφορίες. εγκρίθηκε. Τροπολογία 33, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 34 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα, τροπολογία αριθμός 1 και 10, με 16 μπορούμε να ψηφίσουμε μαζί όλες τις τροπολογίες. 1 και 16 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτονται. Και τώρα ψηφίζουμε την τροποποιημένη γνωμοδότηση ηλεκτρονικά. Ψηφίστε. Πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Ευχαριστούμε. Συνάδελφοι, σκιώδεις, συγητές όλοι, σας ευχαριστούμε πολύ. Επόμενο. ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο το 2016 και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του θέματος. Σόλε. Ε, Η συντάξη γνωμοδότησης είναι ο Ζορδί Σόλε. It's okay. It's okay. It's okay. Καλά το λέω. Ωραία, ευχαριστώ. Συμβαστική πρόταση 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Η ηλεκτρονική επαλήθευση. Έναρξη τη ε, ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 9. Ε, σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 11, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 12, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 13, υπέρ, κατά, αποχές. Νομίζω ότι απορρίπτεται. Παρακαλώ όμως ηλεκτρονική επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία, λήξη τη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 17 υπέρ. Κατά. Αποχές. Παρακαλώ ηλεκτρονική επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 18 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 21 υπέρ. Κατά. Αποχές. Παρακαλώ ηλεκτρονική επαλήθευση της τροπολογίας 21. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. You want to check. Okay. Compromise Η ε, ε, ηλεκτρονική επαλήθευση τη συμβαστικής 4. Έναρξη της ψηφοφορίας, λήξη της ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τροπολογία 23. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 41. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παρακαλώ ηλεκτρονική επαλήθευση της ε, τροπολογίας 41. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 42. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 8 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι εγκρίνεται. Παρακαλώ όμως ηλεκτρονική επαλήθευση. Συμβιβαστική 8 άρχεται η ψηφοφορία, λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 9 υπέρ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 το σημείο 8 της ημερησίας διάταξης ε, είναι το ημερολόγιο για το 2018. Ήδη έχει εγκριθεί από τους ε, συντονιστές και θα θεωρηθεί ότι εγκρίνεται εάν δεν υπάρξει καμία αντίρρηση. Σας ευχαριστώ πολύ, εγκρίνεται. Συνάδελφοι, απομένει μόνο να σας ενημερώσω ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα στα διάφορα και ότι η επόμενη συνεδρία θα πραγματοποιηθεί 21 Νοεμβρίου. Ολοήμερη συνεδρίαση θα είναι. Παρακαλώ. Μην ξεχάσετε ότι θα συμμετάσχουν και μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων που όλοι περιμένουν να συμμετάσχουν ενεργά σε αυτή τη συνεδρίαση. Η Πρόεδρος ευχαριστεί ευγενικά τις Διερμηνείς και εμείς ευχαριστούμε. Ευχαριστεί και τη Γραμματεία. Καλό βράδυ.